Καλώ ε, ε, Καλώς ορίσατε κυρία Τάισεν υποψήφια επίτροπος για απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δεξιότητες και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού η επιστολή του υποψηφίου Προέδρου του κ. Ζαν Κλοντ Γιονκέρ του είπε ότι θα συμβάλλει η κυρία Τάισον να εφαρμόσει συντονισμένα προγράμματα, αυτά που συντονίζονται από τον Αντιπρόεδρο για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας και τον Αντιπρόεδρο για την Ευρώπη και τον κοινωνικό διάλογο. Θα συνεργάζεται στενά με τον Επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων Φορολογήσης και Τελωνίων. Η κυρία Τάισεν θα έχει υπηρεσίες υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Συμπερίληψη, Ένταξη θα την βοηθήσουν όμως και οι εκάτωθοι μονάδες μεταρρυθμίσεως της ε, αγοράς εργασίας, δεξιοτήτων και προσόντων, επαγγελματικής κατάρτισης και πολιτικής για την εκπαίδευση των ελλήκων και δικαιώματων ατόμων με, ειδικές, με αναπηρίες, καθώς και θα επικουρείται και από τη Eurostat. Θα είναι υπεύθυνη και για σχέσεις με τέσσερις υπηρεσίες αρμόδιες για τον τομέα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την υγεία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη πρόθεση επαγγελματική κατάρτιση το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψήφιους επιτρόπους επί τη βάση και παραθέτω γενικών ικανοτήτων, αφοσίωση τον ευρωπαϊκό σκοπό και προσωπική ανεξαρτησία. Θα αξιολογήσει τη γνώση των μελλοντικών τους χαρτοφυλακίων και των διαφόρων ικανοτήτων τους όσον αφορά την επικοινωνία. Πριν την ακρόση να πω ότι έχετε απαντήσει γραπτός, κυρία Τάισον, στα προπαρασκευαστικά ερωτηματολόγια. Οι γραπτές απαντήσεις έχουν διανεμηθεί στα μέλη, σε όλες τις γλώσσες, οπότε είμαστε όλοι καλά προετοιμασμένοι για τις ερωτήσεις που θα σας θέσουμε προφορικά. Κάποια λόγια για την, λόγια για την όλη δομή της ε, συζητήσεως. Η κυρία Τάισον καλείται να κάνει μια αναρκτήρια προφορική δήλωση. Δεν θα είναι μεγαλύτερη από 15 λεπτά. Θα έχει 5 λεπτά στο τέλος της συνεδριάσεως για να ολοκληρώσει την παρουσίασή της. Μετά αυτή την εισαγωγή θα υποβληθούν 45 ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Η συζήτηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με την διαδικασία ping-pong όπως αποκαλείται ο καθένας θα έχει τρία λεπτά στη διάθεσή του μάλλον ένα λεπτό για την ερώτηση δύο λεπτά για την απάντηση τρία λεπτό για την ερωταπάντηση έχουμε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων και γι' αυτό πρέπει να σεβαστείτε σας παρακαλώ ε, με αυστηρότητα το χρονικό όριο θα, θα επιβάλλω τον κανόνα αν ο μιλητής απουσιάζει στο χρόνο που προβλέπεται ότι τεθεί δεν θα υποβληθεί το ερώτημά του, δεν θα υπάρχει διαδικασία catch the eye. Και η Επιτροπή Απασχόληση είναι η καθήλια αρμόδια επιτροπή για την ακρόαση. Αλλά έχουμε και την Επιτροπή Πολιτισμού και την Επιτροπή Γυναικών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση ε, που ασχολούνται, καλύπτουν και αυτές το θέμα. Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους και από αυτές τις δύο επιτροπές και όπως αναφέρεται στον κατάλογο των αγοριτών θα θέσουν διάφορες ερωτήσεις που σχετίζονται με τις εντολές και τις αρμοδιότητες των επιτροπών. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων ανήκει στους συντονιστές και έναν εκπρόσωπο των μη εγγραμμένων μελών. Η διερμηνία ε, παρέχεται σε 23 γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους. Το ίδιο θα κάνω και εγώ σύντομα. Να υπενθυμίσουμε στους ομιλητές ότι αυτό που θα πούν πρέπει να μεταφραστεί μέσω των διερμηνέων. Άρα θα ήταν καλό να μην μιλάμε πολύ γρήγορα. Η κυρία Τάισεν ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την μητρική της γλώσσα, τα Ολλανδικά, για τις απαντήσεις. Το επιχείρημά της είναι ότι θέλει να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται και σαφής. Οι παλαιότεροι συνάδελφοι γνωρίζουν την κυρία Τάισεν, κατέχει ε, πλήρως και την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο ζωντανά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συνεδρίαση και θα μπορείτε να βλέπετε και μαγνητοσκοπήσεις ε, της ακροάσεως στην ίδια στο σελίδα. Θα μιλήσω τώρα τη μητρική μου γλώσσα, σου ειδικά. Θα σας δώσω, θα προβώ σε κάποια αρχικά σχόλια προσωπικής ε, φύσεως που αφορούν την ακρόαση. Ένας Μία από τις ε, πιο έντονες αναμνήσεις από τις εκλογές, ευρωεκλογές φέτο ήταν ένα τηλεφώνημα που έλαβα από έναν ιερέα που εργάζεται για την Σουηδική Εκκλησία, μία ιερέα, στη Νότια ε, Σουηδία, ανησυχούσε πολύ ιερεύς και ήταν απελπισμένη για τη φτώχεια που είδε ε, σε ένα χώρο στάθμευσης ε, στην ε, πόλη της. Έβλεπε σειρά φορτηγών που περίμεναν νέες παραδόσεις και καμιά φορά οι οδηγοί των φορτηγών ζούσαν και ζουν στα φορτηγά, κανείς δεν είχε συλλογική σύμβαση ή κάποια προστασία, δεν πληρωνόταν όταν δεν οδηγούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να πάνε στο σπίτι τους όμως. Περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά την υγιεινή και τα τρόφιμα και όπως ξέρετε ο χειμώνας μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρός στη Σουηδία. Κάποιοι από αυτούς έπρεπε να αποστατευθούν έχοντας ε, μικρές ε, θερμάς, μικρές σόμπες κατασκήνωσης. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατάνε τις μηχανές αναμένες για να ζεσταίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση στον τομέα των μεταφορών και σε πολλούς άλλους τομείς στην Ευρώπη. Είναι κάτι που το βλέπουμε και με γυναίκες εργαζόμενες σε πολλούς τομείς. Αυτή είναι η κατάσταση, η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη όπου τα δικαιώματα των ανθρώπων και όλοι οι κανόνες έχουν θρηματιστεί λόγω της κρίσης και εκείνοι που θέλουν να εργαστούν δεν είναι απλώς άνεργοι, δεν έχουν καν δικαιώματα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πόρα απέχει από τους στόχους της για το 2020. Πάνω από 120 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με φτώχεια κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη. 32,4 εκατομμύρια είναι παιδιά. Ε, τον Ιούλιο φέτος η ανεργία των νέων ήταν στα 22% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις μεταξύ κρατών μελών. Σε κάποιες χώρες είναι τόσο ψηλό το ποσοστό που πάνω από το μισό των νέων της χώρας ε, είναι άνεργοι. Και είδαμε τις συνέπειες αυτού. Το είδαμε και στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών φέτος. Το βλέπουμε όταν βλέπουμε ποιο είναι ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης. Ε, εκφράζεται η απογοήτευση, η απελπισία και απευθύνονται προς αντιδημοκρατικά κόμματα και ακρεφνή κόμματα ε, οι άνθρωποι. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει το 2014 στην Ευρώπη. Σκοπός μας την επόμενη πενταετία είναι να λύσουμε τα προβλήματα της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε νέες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Δεν θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμό σε χαμηλές αμοιβέ και κακές συνθήκες. Ε, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να λύσουμε τα προβλήματα, ο καθένας να έχει τις ίδιες δυνατότητες και να έχουμε ισχυρή αγορά εργασίας. Άρα ε, πρέπει να, πρέπει να κινηθούμε στεναρά. Και ο νέος επίτροπος του τομέα έχει πάρα πολλές ευθύνες για τον χώρο αυτό. Εγώ προσωπικά και οι άλλοι πολίτες της Ευρώπης περιμένουμε η κυρία Τάισεν αρκετά σκληρή και ευφυής, ούτως ώστε να εκτελέσει αυτά τα πολύ σημαντικά καθήκοντα, να είναι αρκετά δυνατή, ούτω ώστε να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές. Είναι, δεν είναι πια η ώρα να καθόμαστε να περιμένουμε, είναι ώρα για δράση τώρα. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τάισεν να κάνει μια εισαγωγική παρέμβαση, να δούμε ποια